Τα πρακτικά της συνεδρίας της 16 Ιουλίου του 2009 να έχει διανεμηθεί. Τα έχετε λάβει και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά αυτά. Δεν βλέπω να υπάρχουν παρατηρήσεις, οπότε τα πρακτικά εγκρίνονται. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έλαβα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Συγγνώμη, μια άλλη πληροφορία θα ήθελα να σας δώσω πρώτα. Οι βελγικές αρχές ε, με ενημέρωσαν για την ανάκληση του κυρίου Ζαν Κλοντ Μπάλκο σε μια θέση που είναι συμβίβαστη με τη θέση του Ευρωβουλευτή με βάση το άρθρο 7 ε, της ε, πράξης για τις καθολικές και άμεσες